Θα ήθελα, συνάδελφοι, να σας ενημερώσω ότι το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και αφορά τις κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινή αυτής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας με βάση το άρθρο 36 της συνθήκης. Όπως βλέπετε η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη μόλις έφτασε και μόλις θα καθίσει θα ήθελα να τη ζητήσω να πάρει το λόγο και να προβεί στη δήλωσή της. Κυρία Μογκερίνη, έχετε το λόγο. Thank you. sorry I was... Uh, Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, έπρεπε να ενημερώσω την Επιτροπή